udgangspunkt, som kommissionen er med, har måske de rigtige Προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι μεν ε, καλύπτει τους, ε, την ορθή στοχοθέτηση, όμως ε, τα σφάλματα εκείνα τα οποία υπήρχαν έγιναν κατανοητά και έγινε προσπάθεια να αλλάξουν αυτά και μάλιστα με επιτυχή τρόπο. Ευχαριστώ. Uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άρης που ανέλαβε τα απλώς κάναμε μια, είχαμε μια μίνι συνέντευξη τύπου ε, με την κυρία Σαμπούνη. Επόμενο ο Θέλω να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος και να προσθέσω ορισμένα στοιχεία διότι δεν ε, νομίζω ότι ε, μόνο για τους διπλωματικούς επισκέπτες από την Επιτροπή αλλά γενικώ και ουσιαστικά είναι καλό να υπάρχουν τέτοιες ε, πρωτοβουλίες που να εξετάζουν την ευελιξία των κρατών μελών και την νομιμότητα της νομοθετικής διαδικασίας διότι στο Κοινοβούλιο πρέπει να κάνουμε συμβιβασία. Πρέπει να προσεγγίσουμε τους άλλους και ε, είμαι πολύ, αμφιβάλλω πάρα πολύ για τις διεργασίες αυτές. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λεχθεί, διότι δεν ξέρω αν οι καταναλωτές κατά τη στιγμή που αγοράζουν κάτι σκέφτονται τα δικαιώματά τους. Υποθέτω δηλαδή, ε, εγώ ζω στα σύνορα της Γαλλίας και πηγαίνω σε ένα μεγάλο κατάστημα πέρα από τα σύνορα και ε, πηγαίνω εκεί διότι από θέμα εμπιστοσύνης και οικονομικά θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σημείο και ε, ως επτοπλίστων ε, τα πράγματα έχουν σήμανση γαλλική. Ε, οπότε εμείς ρωτάμε εάν ο καταναλωτής ξέρει τα δικαιώματά του. Αλλά εγώ στη ζωή μου πρέπει να πω ότι ποτέ δεν σκέφτηκα όταν πηγαίνω να αγοράσω στη Γαλλία πράγματα των οποίων δεν αντιλαμβάνουμε τη σήμανση και ε, ε, ε, στο κατάστημα αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί με γερμανικές πινακίδες και αγοράζουν συλλήβδιν εκεί οπότε ίσως η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Λοιπόν, επιπλέον θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατή να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση διότι υπάρχει και το ενοχικό δίκαιο και πρέπει να δούμε ε, ε, πότε υπάρχουν προθεσμίες για τη λήξη της ισχύω. Έχουμε δηλαδή πολλές πληροφορίες, αλλά ε, πρέπει να εξετάσουμε εάν υπάρχουν νομικές συνέπειες, εάν οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις. Και αυτή η αντιμετώπιση είναι διαφορετική στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχουν ε, ε, σημαντικές ε, επιπτώσεις νομικές για παραβιάσεις της πληροφόρησης μπορεί κανείς να κρατήσει τον πύχη πολύ ψηλό και όπου υπάρχουν πιο περιοριστικές επιπτώσεις τότε ο πύχης είναι πολύ πιο χαμηλός. Είναι θέματα δηλαδή που πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και πρέπει να σκεφτούμε σύμφωνα με την απόφαση την οποία πήραμε για την πράσινη βίβλο ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και εις ε, ε, βαθμιαία και εις ε, το, τα θέματα τα νομικά, διότι είχαμε συμφωνήσει ότι σε θέματα όπως οι ορισμοί για τον καταναλώτη, για τις προθεσμίες λήξεως, θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίες διατάξεις για όλες τις οδηγίες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο. Βλέπω όμως ότι συμβαίνει το αντίθετο, διότι όσον αφορά το θέμα της εναρμόνισης δεν πρέπει να βασιστούμε στον κατώτατο παρανομαστή. Θα πρέπει ορισμένα θέματα να εμβαθυνθούν, να δούμε τι είναι σημαντικό και τι, είναι, και τι όχι. Πρέπει όμως να σας πω ότι εδώ δεν θέλουμε να αποβλέπουμε σε μία κατώτατη εναρμόνιση, αλλά θα θέλαμε να εξετάσουμε και ποιο είναι το ανώτατο όριο εναρμόνισης κατά τρόπον ώστε ε, να υπάρχει μία, ε, ε, ένας καθορισμός των ορίων αυτής της εναρμόνισης. Διαφορετικά το κάθε κράτος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ενώ εμείς, ο ένας μπορεί να πει ότι εμείς θα να βάλουμε κατώτατο επίπεδο δύο χρόνια και όχι περισσότερο από τόσα χρόνια. Δηλαδή μπορεί κανείς να βάλει ένα κατώτατο και ένα ανώτατο όριο, να υπάρχει μία ευελιξία αλλά να είναι οριοθετημένη κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία εναρμόνιση. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια μεγάλη πίεση που δεν έχει αναφερθεί σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, διότι μέχρι τώρα όλες αυτές οι οδηγίες δεν αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών αντιλαμβάνομαι την ε, θέση της, πολιτικής, ε, Ευρωπαϊκής ε, ε, ε, Επιτροπής, η οποία λέει ας προχωρήσουμε με αυτά τώρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι ε, εάν περιλάβουμε και την παροχή υπηρεσιών θα υπάρξουν ε, ιδιαίτερες επιπτώσεις και ε, ίσως θα έπρεπε να εξαιρέσει κανείς αυτό το θέμα και να το ρυθμίσει χωριστά. Αυτές είναι οι πρώτες μου ιδέες και για να επαναλάβω η νομοθετική εργασία κατ' εμέ, ε, όταν ε, την εξετάζω και βλέπω και τις συνήθειες ε, και στο Συμβούλιο, ε, βλέπω ότι έχει δικές του θέσεις όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και ε, θα έπρεπε τα θέματα αυτά να προωθηθούν και για άλλα θέματα ο πολίτης ε, θα εξυπηρετηθεί καλύτερα εάν καθυστερήσουμε και αφήσουμε για τους επόμενους νομοθέτες να έχουν κάτι να κάνουν και αυτοί. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πριν περάσουμε στον κατάλογο των ομιλητών. Να καλωσορίσω την κυρία Μάινε, την κυρία Μπαμόντι από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Θα τους δώσω την ευκαιρία να σχολιάσουν ε, μετά την εκτενή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας για να μας πούνε την δική τους οπτική γωνιά, να σχολιάσουν λίγο αυτό που θα ακούσουν να σας ενημερώσω ότι είχαμε μια λεπτομερή ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Σαμπούνη για τα θέματα των δικαιωμάτων καταναλωτών και μετά, ε, τώρα εμείς συνεχίζουμε αυτή τη γενική συζήτηση. Λοιπόν, η κυρία Γκέπχαρτ και η κυρία Ρόιτεβερ, τον κύριο Κότζισνικ και τον κύριο Μπαρνιέ. Αλλά και αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο, κανένα πρόβλημα. Κάποιος άλλος ήθελε να πει κάτι και ο κύριος Βιγιόν. Ας ξεκινήσουμε και... Δεν βλέπω καλά μέχρι εκεί. στην πράσινη κάρτα εκεί. Εντάξει, θα σας... Ε, θα σημειώσω με το όνομα. Λοιπόν, η κυρία Γκέπχαρτ. Yeah, Ευχαριστώ πολύ, Μάκομ. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα οποία πιο πριν είχα προναφέρει. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λέχνερ πρώτα για το γεγονό ότι μας κατέδειξε. Δεν ξέρω αν εν ονόματι του ιδίου ή εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής του ομάδας ότι στην απόφαση, θεμελιώδη απόφαση που ελήφθη ήδη στην Ευρωβουλή ότι δηλαδή δεν επιθυμούμε πλήρη εναρμονισμό αλλά μια μεικτή προσέγγιση για τον εναρμονισμό αν αυτό δηλαδή θέλουμε, ότι αυτό θέλουμε να συνεχιστεί. Με αυτή τη βάση νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και έτσι πολλά μπορούμε να αποφύγουμε όσον αφορά τριβές μεταξύ κοινοβουλευτικών ομάδων διότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Υπήρξε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μακρόχρονα συζητήσαμε προτού λάβουμε αυτή την τελική μας απόφαση. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω και θα ήθελα εδώ να επικεντρωθώ σε αυτό το σημείο που ο κύριος Λέχνερ προανέφερε, δηλαδή τον βαθμό εναρμονισμού ή τι σημαίνει ο πλήρης εναρμονισμός ή τι δεν σημαίνει αυτός. Νομίζω αυτό το οποίο προτάθηκε, δηλαδή μία βήμα προς βήμα προσέγγιση προς τα εμπρός είναι η ορθή προσέγγιση. Είναι και η προσέγγιση που εμείς ως σοσιαλδημοκράτες, γυναίκες και άνδρες ακολουθούσαμε πάντα σταδιακά βελτιώσεις, βήμα προς βήμα εναρμονισμός, όχι εξάπαντος δια μιας ε, εναρμονισμός. Νομίζω αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης, βήμα προς βήμα. Και αυτό ανταποκρίνεται και στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στο άρθρο 153, αν θυμάμαι σωστά όσον αφορά τον αριθμό του, αναφέρεται σαφώς ότι κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να υιοθετήσει περαιτέρω νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται ανταποκρίνεται και συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό είναι και αυτό κάτι που πρέπει να σεβαστούμε, δηλαδή όσον αφορά τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να γίνει σεβαστό. Το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει φυσικά να προβληματιστούμε και να δούμε τι σημαίνει πλήρης εναρμονισμός. Ας υποθέσουμε ότι θα κάναμε κάτι τέτοιο. Ας υποθέσουμε ότι θα ακολουθούσαμε την οδό του πλήρους εναρμονισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα είχαμε το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων προστασίας καταναλωτών σε όλες τις χώρες. Αυτό καταδείχθηκε σαφέστατα όταν είχαμε την ακρόαση που διεξαγάγαμε. Και σε μία από τις ερωτήσεις προς την κυρία Μπαρόλο Βασέλ που τότε ως αρμόδια επιστήμων είχε παραστεί, όταν της τέθη αυτό το ερώτημα, τον κύριο Σβάμπ κατά τα άλλα, έτσι, και πρόκειται για την αγορά αυτοκινήτου με προσυμβάσεις προ, ε, όπου ο κύριος Σβάμπ είπε ότι στη Βάδη Βίρτεμβέργη υπάρχουν πολλοί Γάλλοι που κάνουν τέτοια προσυμβόλαια και εκινήσατε από την υπόθεση κύριε Σβάμπ ότι το δίκαιο στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι διαφορετικό είπατε. Επειδή οι Γάλλοι αγοραστέ, δηλαδή οι Γάλλοι καταναλωτέ, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να υπαναχωρήσουν από τέτοια προσυμβόλαια, προσυμβάσει και ότι δεν θα ήταν υποχρεωτικό ο σεβασμός τους. Και εσείς είχατε καταλήξει στο συμπέρασμα υπάρχει διαφορετικό δίκαιο στη Γαλλία και στη Γερμανία. Και η κυρία Μπέντε Μασέλ είπε ότι όχι, δεν αληθεύει λέει αυτό. Στη Γαλλία ισχύει απόλυτα το ίδιο δίκαιο όπως στην Γερμανία. Προσύμφωνα είναι προσύμφωνα και πρέπει να είναι σεβαστά. Στη Γαλλία, μέσω όμως μιας διαφορετικής παράδοσης ε, και ε, πολιτισμού αυτής της παράδοσης υπάρχει συνένεση συνενετική αντιμετώπιση. Δεν βρίσκω τώρα τον όρο, πώς να το πω για την ας το πω γενεοδορία ή την, ε, ε, το ευρύτερο πλαίσιο που θα ισχύει όπου οι Γάλλοι πολιτές λένε αν δεν θέλετε εσείς να αγοράσετε αυτό το αυτοκίνητο τότε δεν θα ισχύει το προσύμφωνο. Αυτό είναι γενεοδορία, δεν είναι δίκαιο. Στη Γερμανία όμως δεν υπάρχει αυτή η γενεοδορία αντιμετώπιση. Το προσύμφωνο ισχύει ως προσύμφωνο. Ακόμα και αν ίσχυαν λοιπόν τα ίδια δικαιώματα υπάρχει διαφορετική παράδοση για την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων στα ε, νομικά μας συστήματα προβλήματα. Και γι' αυτό δεν έχει μεγάλο νόημα να θέλουμε να αντιπαρατεθούμε για αυτό το θέμα και να πούμε θα κάνουμε ένα κοινό δίκαιο, ε, ε, πλαίσιο δικαιωμάτων και αυτό θα δίνει ένα κοινό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο με επηρέασε περαιτέρω στον προβληματισμό μου και στις σκέψεις μου και με ενίσχυσε στο να πω θα παραμείνουμε σε αυτή την προσέγγιση της μικτής ρύθμισης, του, μικ, του μικτού εναρμονισμού. Και θα πρέπει να δούμε τώρα πού έχει νόημα, πού έχει νόημα να υπάρξει εναρμονισμός στον, ε, στον ορισμό του καταναλωτή, για παράδειγμα, των καταναλωτών ή ε, για παράδειγμα του δικτύου παρόχης ή για τον ορισμό όταν έχουμε περιόδους προθεσμίες για την ανάκληση κάποιων ε, υποχρεώσεων, ε, κάποιες ημέρες ή εβδομάδες, να πούμε ότι για όλους τους τομείς θα ισχύει η ίδια προθεσμία. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάποιο εναρμονισμό, αλλά εδώ και για το δικαίωμα ανάκλησης, όπου πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις υπάρχουν, πρέπει να προβληματιστούμε, να δούμε μπορούμε να το κάνουμε αυτό ή όχι. Δεν θα έπρεπε να σεβαστούμε ότι υπάρχουν, υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις στα κράτη-μέλη μας. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση θα έλεγα. Να λάβουμε υπόψη και να σεβόμαστε αυτές τις διαφορές όταν προσεγγίζουμε το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήθελα να ενισχύσω και να εντείνω σε σχέση με τις εξαιρέσεις ε, που είχαν ληφθεί στο, έγιναν στο παρελθόν. να η κυρία Βόητε και μετά ο κύριο Κοζιδέσκο Μπαγνιέ, and uh, Mr. κύριος Πουπάκης και κύριος Σβάμπ. Α, και κυρία Βάιλερ. Η κυρία Βάιλερ και μετά ο κύριος Σβάμπ, γιατί είχατε σηκώσει το χέρι σας νωρίτερα. Α, κι άλλος ένας ομιλητής. Λοιπόν, εδώ κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Γιατί μέχρι τις 12 πρέπει να τελειώσουμε με αυτό το θέμα κυρία Ρόιτεμπεργκ. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ ότι καθυστερούμε πολύ σε αυτή τις συζητήσεις. Δύο μήνες τραβάνε οι συζητήσεις μέχρι τώρα και θα, έχουν, θα κρατήσουν και άλλους, και άλλους δύο μήνες τουλάχιστον. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια πολιτική συμφωνία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι... Αυτό είναι, το, είναι ο στόχος μας. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και από όλες τις συζητήσεις που έχουμε που είχαμε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι έχουμε μπλέξει τα πράγματα. και θα πρέπει η Επιτροπή, η Κομισιόν, να παίξει έναν ηγετικό ρόλο. Ακούγονται διάφορα θέματα, υπάρχουν ε, ε, διαφορετικές διατάξεις σε διαφορετικές χώρες, ε, μας λείπουν πληροφορίες, μας λείπουν γνώσεις. Και θα πρέπει να μας διαφωτίσει η Κομισιόν, να ξέρουμε και τι ισχύει όσον αφορά το δίκαιο των καταναλωτών στις διάφορες χώρες. Γι' αυτό απευθύνομαι προς την Κομισιό να μας δώσει λεπτομερείς πληροφορίες, να μας δώσει μια εικόνα, αν θέλετε, των όσων συμβαίνουν στις διάφορες χώρες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, αλλά τέλος πάντων έναν πίνακα να δούμε. Αυτές οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούν να καλυφθούν. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλουμε να επηρεάσουμε την, τις εμπορικές πολιτικές των κρατών μελών ε, σε εσωτερικό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι αναγνωρίζω ότι ενδεχόμενα να υπάρχει μια κάποια προστιθέμενη αξία όσον αφορά ας πούμε την παράταση της εγγύησης. Αυτή όμως η παράταση της εγγύησης δεν επηρεάζει αυτή καθεαυτή την ποιότητα του προϊόντος. Λοιπόν, αυτό αυτή, αυτός, αυτή η διάταξη που αφορά την περίοδο εγγύησης χρειάζεται να εναρμονιστεί ή όχι. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πνίξουμε και τις, ε, με υποχρεώσεις τις διάφορες επιχειρήσεις. Γι' αυτό Πάλι απευθύνομαι στην Κομισιόν και ρωτώ γιατί πρέπει να έχουμε την μέγιστη εναρμόνιση σε σχέση με την ελάχιστη. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της μέγιστης εναρμόνισης. Διότι εγώ καταρχάς συμφωνώ με την Κομισιόν. Θέλουμε να ε, ενδυναμώσουμε τις ε, διεθνείς συναλλαγές, τις συναλλαγές μέσω του ίντερνετ και για να γίνουν όλα αυτά πρέπει οι διατάξεις να είναι ξεκάθαρες. Πρέπει οι καταναλωτές να ε, ξέρουν τα δικαιώματά τους, πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν τους, τις διάφορες διατάξεις που ισχύουν, οι ορισμοί να είναι σαφείς και κατανοητοί γιατί στο κάτω-κάτω εμεί είμαστε υπεύθυνοι για την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω τώρα τον κύριο Κοσνίσκι, που είναι ένα νέο μέλο τη Επιτροπή μα. <laughs> Και νομίζω ότι είναι το, το μόνο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έρχεται με το ποδήλατο από την εκλογική του περιφέρεια ε, μέχρι, μέχρι εδώ ε, ως δέσμευση που ανέλαβε έναντι των ψηφοφόρων του. Πρόεδρε, θα μιλήσω τσέχικα. Πρόεδρε, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της Κομισιόν. Θα ήθελα να χαιρετήσω και τους ε, συνεργάτες ε, των ε, βουλευτών και τους διερμηνείς. Τέλος πάντων, να καλωσορίσω όλους, μια και είμαι καινούριο εδώ. Ήθελα να πω ότι ναι, μπορεί να είμαι καινούριο εδώ, αλλά ασχολούμαι εδώ και μερικά χρόνια με θέματα που άπτονται της βελτίωσης και της απλούσευσης της νομοθεσίας. Τώρα, σχετικά με το θέμα που μας απασχολεί, την προστασία των καταναλωτών. Καταρχάς να πω ότι η Κομισιό έχει κάνει πολλή δουλειά και όσον αφορά την απλούστευση της νομοθεσίας και όσον αφορά τον κατακαιρματισμό, αν θέλετε, ε, των θεμάτων. Ε, διότι θα πρέπει να ξεμπλέξουμε καταρχάς τα, τα θέματα και για κάθε θέμα να υπάρχει μια νομοθεσία. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρη συναρμόνιση. Άλλοι συνάδελφοι έχουν διαφορετική άποψη. Μέχρι στιγμής στην προστασία των καταναλωτών εφαρμόζουμε την αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να διατηρήσουν ή μπορούν να διατηρήσουν πιο αυστηρές διατάξεις. Όμως θεωρώ ότι στις ε, ενδοκινοτικές συναλλαγές αυτό είχε αρνητικά, αρνητικές επιπτώσεις, διότι υπήρχαν ε, επιχειρήσεις που δεν ε, ήθελαν να πουλήσουν σε άλλες χώρες ε, ή δεν μπορούσαν και αυτό νομίζω ότι ήταν εις βάρος του, εμπορίου. Η Κομισιό προσπαθεί να πετύχει καλύτερη, καλύτερες συναλλαγές, μια πιο εύρυθμη λειτουργία της ιστορικής αγοράς. Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Α, χάσαμε λίγο το κατάλογο. Α, ο κύριος Μπαγνιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις για ένα κείμενο το οποίο είναι σημαντικό και περίπλοκο. Και δεν, δεν θα ήθελα να επαναλάβω ερωτήσεις που έκαναν άλλοι συνάδελφοι και πάνω στις οποίες ε, χρειαζόμαστε ε, τα φώτα των συναδέλφων, της Κομισιόν κυρίως και της Προεδρίας. Το κείμενο αυτό είναι σημαντικό, το ξέρουμε όλοι, για να διευκολύνουμε την ε, εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και είναι σημαντικό επίσης για να διασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην μέγιστη προστασία των καταναλωτών αφενός και να ε, περιορίσουμε τον κίνδυνο ε, που, και, και το βάρος που αντιπροσωπεύουν 27 ε, διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες για τις επιχειρήσεις. Τα καταλαβαίνω τις δυσκολίες που θέτει αυτό το κείμενο γιατί μπορεί κάποια κρατημέλη τα οποία θα ήθελαν δεν θα μπορέσουν να υιοθετήσουν μέτρα πιο προστατευτικά για τους καταναλωτές για κάποιους τομείς. Αυτός είναι ένας κίνδυνος ο οποίος υφίσταται και αυτό αυτή, αυτή είναι μια διευκρίνηση που θα ήθελα να μου δώσουν οι συνάδελφοι. Επίσης ε, άκουσα ότι οι επαγγελματίες ε, θα έχουν ε, δυσκολίες να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής και πώς συνδέεται και πώς επηρεάζεται η η οδηγία αυτή με τα άλλα υπάρχοντα νομοθετικά κείμενα. Και εδώ χρειαζόμαστε τα φώτα της Κομισιόν. Επίσης, κάποια άλλη διευκρίνηση την οποία θα ήθελα είναι ε, η συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν την μέγιστη και την πλήρη εναρμόνιση και αυτούς που θέλουν μια μέγιστη εναρμόνιση αλλά συγκεκριμένα εστιασμένη εναρμόνιση. Η Κομισιόν θέλει αυτή την μέγιστη εναρμόνιση που και που δημιουργεί κάποια προβλήματα, τα οποία προσπάθησα να αναφέρω προηγουμένως. Πιστεύω ότι πρόσφατα η Κομισιό έχει κάπως εξελιχθεί, δηλαδή έχει προχωρήσει τις, ε, τις σκέψεις και προχωράει σε μια εναρμόνιση εστιασμένη. Αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσει η Κομισιό. Το κατάλαβα καλά ή όχι. Και όταν λέμε ε, εστιασμένη εναρμόνιση, σε ποιους τομείς εστιάζει την εναρμόνιση. Και θα ήθελα και την άποψη της Προεδρίας από του τους. Uh, Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και ένα άλλο νέο μέλος, τον κύριο Ποπάκη. Ευχαριστώ. Σαν νέος Ευρωβουλευτής θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τη χαρά μου που συμμετέχω στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία Καταναλωτών, γιατί και προάγει την ενοποίηση Ευρώπης Ευρώπη μέσω της ενιαίας αγοράς αλλά και συμβάλλει στο κοινωνικό συνολό προωθώντα τα συμφέροντα των καταναλωτών που μα ενδιαφέρει. Αναφορικά με την οδηγία θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι ο σκοπός της πρότασης είναι πραγματικά η δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Καθώς απλωστεύονται κανόνες ε, για τα 27 κράτη-μέλη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών κατά την πρόσβασή του σε αγαθά και υπηρεσίε. Θα πρέπει όμω να επισημάνω και εγώ, όπω και άλλοι προηγούμενα από μένα, συνάδελφοι, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εφόσον πρόκειται για πλήρη εναρμόνιση. Για να μην υποβαθμιστεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που έχει επιτευχθεί ε, σε συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες εθνικές διατάξεις. Παράδειγμα, στη χώρα μου, την Ελλάδα, το κύμα της πρότασης, όπως έχει κατατεθεί από την Επιτροπή, μειώνει το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με ισχύοντα το εθνικό μας δίκαιο να αναφέρω ενδεικτικά δύο-τρει περιπτώσει. Δεν γίνεται αναφορά σε υποχρέωση συντήρηση, επισκευή και επάρκεια ανταλλακτικών για, την για όλη πιθανή τη διάρκεια ζωή προϊόντο. Περιορίζεται η άσκηση δικαιωμάτων των καταναλωτή σε περίπτωση έλλειψη συμμόρφωση του εμπόρου. Δεν γίνεται πρόληψη για δυνατότητα προσωρινή αντικατάσταση του αγαθού σε περίπτωση υπέρβαση 15 μέρου και αρκετά άλλα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν οι επιπτώσει που θα έχει η εν λόγω πρόταση στην πράξη και ο αντίκτυπος στα υφιστάμενα δικαιώματα και μέσα ένομης προστασίας, καθώς και στην ισορροπία με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Δίκαιο. Διαβάζοντα το έγγραφο τη εργασία που συνέταξε η προηγούμενη Επιτροπή Ιστορική Αγορά, πιστεύω ότι θα ήταν καλό να κινηθούμε σε αυτή τη βάση, καθώ πολλοί από αυτού του προβληματισμού τίθενται, αλλά να διασφαλιστούν οι ευνοϊκότερε διατάξει σε κάθε χώρα για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Διγιό είναι ο Βιγιό είναι επόμενος και μετά η κυρία Βάιλερ και θα έδινα τον τελευταίο λόγο στον κύριο Σουάμπ. οπότε αντιλαμβάνουμε ότι ανάμεσά τους θα μπει και ο κύριος Τσεσκόφσκι. Ο κύριος Βιγιό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι είναι ίσως ε, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο πολιτικά θέματα στην ημερήσια διάταξή μας και θα ήθελα να σας πω ότι στην Ολλανδία στην προεκλογική περίοδο τα δικαιώματα των καταναλωτών συζητήθηκαν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ καλή φήμη όσον αφορά τα ε, δικαιώματα του καταναλωτού και έχει βελτιωθεί η κατάσταση ε, στα διάφορα κράτη λόγω των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η ιδέα λοιπόν αυτής της πλήρους εναρμονήσεως θεωρείται από τη χώρα μου ένα πρόβλημα το οποίο ίσως χαλάσει την εικόνα που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ιδίω όσον αφορά στις ε, εγγυήσεις και στη διάρκεια τους υπάρχουν προβλήματα. Τα δύο χρόνια είναι λιγότερο από αυτό που υπάρχει για προϊόντα με μακριά διάρκεια ζωής και δεν είναι δυνατόν οι Βρυξέλλες ε, αντί να βελτιώνει να μειώνει τα δικαιώματα δικαιώματα του καταναλωτού. Είναι λοιπόν βασικό να συμπληρώσουμε όπως ε, είπαν πολλοί ότι ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται προς όφελος του καταναλωτού και όχι να μειώνει τα δικαιώματα που έχει. Διάβασα το έγγραφο εργασίας με μεγάλο ενδιαφέρον και βλέπω ότι πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο και το Μάιο και συμπληρώνει με χρήσιμες ιδέες να σεβόμαστε τις ε, επιχειρήσεις, να υπάρχουν ενιαία δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν λάβουμε υπόψη την εικόνα που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να είναι σύμμαχός τους και όχι να μειώνουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει το έργο της εναρμονήσεως να χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν ξέρω αν είναι προς όφελος ε, των επιχειρήσεων να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και η ισορροπία δεν είναι να μειώσει κανείς ε, την ε, εναρμόνιση αλλά να δούμε ποια είναι η ισχύουσα κατάσταση, ποια είναι τα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο. Δεν θέλω να μιλήσω για μερικά μέτρα αλλά πώς μπορούμε να έχουμε ε, παρεμφερείς ρυθμίσεις και πού πρέπει να δεχτούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον υπάρχουν εθνικές διαφορές οι οποίες σιγά σιγά θα μπορέσουν ε, να ε, προχωρήσουν και πάντοτε πρέπει να είναι προσόφερος του καταναλωτή. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας δώσει ένα κατάλογο για τις ε, πρακτικές προτάσεις σε σχέση με την εθνική νομοθεσία και στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για πλήρη εναρμόνιση ή υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάιλερ τώρα. αστιν Λοιπόν, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία έχω πει εγώ στο παρελθόν, ούτε αυτά που είπαν και οι άλλοι, παρόλο που διαφέρει η άποψή μου διότι όλοι έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση, πράγμα που αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει μόνο προς τα έξω αλλά και προς το Κοινοβούλιο να μπορέσει να πείσει γιατί έχει διατυπώσει αυτή την πρόταση με αυτόν τον τρόπο. Άκουσαμε με τα μεγάλη προσοχή γιατί ο κύριος Λέχνερ θεωρεί ότι είναι περιττή τέτοια ρύθμιση και συμφωνώ διότι ότι αναφέρομαι ότι ουσιαστικά ε, πρόκειται για τις ε, παραμεθόριες περιοχές και όχι για τον καταναλωτή που πάει να ψωνίσει στη γωνία. Ε, υπάρχουν ε, πλήρεις εναρμονήσεις σε άλλα θέματα ανταγωνιστικότητος τα οποία λειτουργούν καλά αλλά τώρα υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το οποίο οι περισσότεροι είναι αντίθετη. Είναι ίσως πρόωρο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το θέμα αυτό. Κάνω όμως μία έκκληση προς τους συναδέλφους. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό να πούμε ότι στα 26 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από, μάλλον όχι λάθος, από τα 27 κράτη-μέλη σε 26 κράτη-μέλη υπάρχει μία μείωση της προστασίας των καταναλωτών εάν υιοθετηθεί αυτή η οδηγία. Θεωρώ ότι αυτό είναι υπερβολή. Δηλαδή δεν συνάδει με τις πραγματικές έρευνες που έχουν γίνει και ότι όλοι οι φόβοι που έχουν εκφραστεί θα οδηγήσουν σε ε, ένα χειρότερο δίκαιο για τους καταναλωτές. Και επίσης αμφισβητώ ότι είναι ε, ε, ένα μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις όπως είπε διάφοροι συνάδελφοι, η κυρία Ρότοβα και άλλους. Δηλαδή δεν θα πρέπει όλα να είναι ευθυγραμμισμένα. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές και λόγω παραδόσεων διότι ο έμπορος μου στη γωνία του σπιτιού μου μου επιτρέπει να αποχωρήσω από ένα προσύμφωνο πράγμα όμως ε, το οποίο δεν μπορώ να απαιτήσω για το γείτονά μου αυτό το κάνει για το δικό μου το χατήρι και θα μείνει έτσι ε, και θα εξασφαλίζεται και στο μέλλον άρα η προσωπική επαφή με τον έμπορο με, ε, τον, με τη γειτονιά είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ε, οι σχέσεις μέσω του διαδικτύου που έχει, ε, όπου υπάρχει ανωνυμία και όπου υπάρχουν ε, και οι περισσότερες καταχρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα θα μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι της απόψεως ότι όντως θεωρεί ότι η πρόταση αυτή είναι μία βελτίωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα, από όλα τα σχόλια. Νόμιζα ότι όλοι είναι αρκετά ε, αμφίβολοι γι' αυτό. Τώρα λοιπόν θα καλέσω ένα άλλο νέο μέλος της Επιτροπής μας και μετά ο κύριος Σβάμπα θα κλείσει, θα είναι ο τελικός ομιλητής. ο κύριος Τρεσκόφσκι. Ελπίζω να έχω προφέρει σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνατε να ε, ε, προφέρετε το όνομά μου. Θέλω να αναφερθώ εις ε, τα μέτρα για την αποκατάσταση. Ε, ε, τα γιατρικά δηλαδή, διότι ένα στοιχείο της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, αν το δικαίωμα επιλογής πρέπει να το έχει ο έμπορος ή ο καταναλωτής και νομίζω ότι πολλοί αγοράζουμε κάτι το οποίο αγαπάμε και μετά από την πρώτη επισκευή αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε και στην τρίτη επισκευή ε, αρχίζουμε να μισούμε και το προϊόν και τον κατασκευαστή του. Ίσως λοιπόν πρέπει να ρωτήσουμε αν έχει γίνει μία, μία μελέτη επιπτώσεων για να δούμε αν θα πρέπει να υπάρχει, να, να βαρύνει πλάστιγκα προς τον καταναλωτή και αν αυτό θα συνεπέχεται περισσότερα έξοδα. Και τώρα ο κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τη συζήτηση ιδίω με τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου ο, την παρακολούσαμε πολύ ενδιαφέρον και τη βρήκα πολύ σαφή ιδίω όσον αφορά την, τα σχόλια του κυρίου Κόσεβικ από την Τσεχία ε, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ήρθε με το ποδήλατο από, έως τις Βρυξέλλες και υποθέτω ότι δεν τα πράγματα του θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ε, μία διαφορά απόψεων όχι μεταξύ ε, της βιομηχανίας και ε, του καταναλωτή απλούστατα πρέπει να δούμε θέλουμε να υπάρχει μία ευρεία επιλογή για τον καταναλωτή ή μεγαλύτερη προστασία. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μία ισορροπία που να επιτρέπει ένα σωστό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Σε ορισμένα κράτη ε, η αυστηρή νομοθεσία δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυστηρή προστασία του καταναλωτή ή συμφέρουσες τιμές. Ίσως όπως είπε η κυρία Βάιλερ μπορεί η κατάσταση να είναι τελείως διαφορετική. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή και ε, στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο εναρμόνισης και γι' αυτό πολύ σωστά είπε ο κύριος Μπαρνιέ ότι το ερώτημα είναι πόσοι συμφωνούν να υπάρξει μια ευρεία εναρμόνιση δηλαδή πόση συνένεση υπάρχει για αυτόν τον στόχο ελέγχθη ότι πρέπει να δούμε ποια είναι τα δικαιώματα του κρατούς μέλους για την, ε, ε, για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτού αλλά πρέπει να δούμε και ε, ποια είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα δικαιώματα του καταναλωτή και της επιχειρήσεως και να μπορέσουμε να τα ισοσκελίσουμε και να κάνουμε μία προσπάθεια ενίας αντιμετωπίσης Ελπίζω όμως ότι υπάρχει μία προσπάθεια προσεγγίσεως του δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τα εμπορεύματα, τα οποία θέλει κάποιος κατανοητής να αγοράσει ενδεχομένως και εκτός της δικιάς του πατρίδας και όπου θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες νομικές διατάξεις οι οποίες θα βελτιώσουν το αγοραστικό αυτό πλαίσιο. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η συζήτηση σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντική και κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα αλλά ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία Σαμπούνη. Εάν όντως το θέμα αυτό πρέπει να προβληθεί και στην κοινή γνώμη θα πρέπει να δώσουμε σαφή παραδείγματα τα οποία ακόμη δεν έχουμε ακούσει. Και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπον ώστε να είναι αποδεκτό από την πλειοψηφία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και για να μπορέσουμε στο μέλλον να αποδείξουμε την ποικιλομορφία της εσωτερικής αγοράς ε, για να ενισχύσουμε και τους μικρούς εμπόρους και να έχουμε λιγότερα ε, McDonald's ε, και Burger King και περισσότερα μικρά καταστήματα, πράγμα το οποίο θα ήταν μεγάλο προσόν για την εσωτερική αγορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε ουσιαστικά στοιχεία και ελπίζω ότι αυτά θα μπορέσει να μου τα διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ήταν ε, πολύ καλή συζήτηση με πλούσια συμμετοχή και επιχειρηματολογία από όλους σας και ε, νομίζω ότι εμπλουτίσατε την πρόταση. Θα κάνω ορισμένα σχόλια σχετικά με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας στο τέλος, αλλά τώρα θα ήθελα και πάλι να, να καλωσορίσω την κυρία Μπερμόντι, ε, μάλλον όχι, την κυρία Μάινερ, η οποία θα μιλήσει. Όποιο και από του δύο είναι θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πούνε διότι έχουν εμπλακεί πολύ σε αυτή τη συζήτηση. Ίσως δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε σε όλα τα θέματα και όλες τις ερωτήσεις αλλά θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες όταν θα καθοριστεί ένα συζητητή. Άρα σας δίδω τώρα τον λόγο για να σχολιάσετε ό,τι ελέγχθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να προλογίσω λέγοντας, είναι μεγάλη χαρά να σας βλέπω στην έδρα του Προέδρου και σας συγχαίρω για την εκλογή σας στο αξίωμα αυτό. Συνεργαστήκαμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για αρκετά θέματα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και για αυτό το θέμα στο μέλλον. Η πρόταση αυτή και αυτό ο χαρτοφύλακα το χαρτοφυλάκιο πάνε στον πυρήνα, στην ουσία των αρμοδιοτήτων των μελών αυτής τη κοινοβουλευτική Επιτροπής, αν επιτρέπετε να το πω αυτό, διότι αφορά όχι μόνο την πολιτική για του καταναλωτέ, παρότι είναι μια πρόταση μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων από πλευρά τη Επίτροπή του Αρμοδίου Επιτροπού, όπως αφορά και, όπω ανέφεραν και αρκετοί προλαλήσαντε, και σε ένα άλλο θέμα, <clears throat> στην ίδια την ενιαία εσωτερική αγορά. Και γι' αυτόν τον λόγο με εντυπωσίασαν οι παρατηρήσεις του, της κυρίας Ρόιτροβα, του κυρίου Κουσέφνιες και οι τελικές παρατηρήσεις του προλαλήσαντος κυρίου Σβάμπ. Η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντάσσοντας αυτήν την πρόταση ήταν να καταφέρει να πετύχει μια πραγματική ας το πω έτσι, ένα ε, εφικτό επίπεδο της ενιαίας εσωτερικής αγορά σε όλα τις λεπτομέρειες. Όλα τα στοιχεία που είχαμε στη διαθέσή μας έδειχναν ότι αυτή η ενιαία εσωτερική αγορά δεν υφίσταται ακόμα. Πολύ λίγοι καταναλωτές συνειδητά αγοράζουν διασυνοριακά σήμερα. Αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες που τους παρέχονται όταν ταξιδεύουν επαγγελματικά ή για λόγους αναψυχής. Αλλά δεν είναι πολλοί εκείνοι που συνειδητά επιλέγουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρει η εσωτερική αγορά για την επιλογή από ένα ευρύτερο εύρος αγαθών ή επιλογή αγαθών σε χαμηλότερες τιμές και έχουμε τεκμήρια και αποδείξεις ότι υπάρχουν αυτές οι χαμηλότερες τιμές αυτών των αγαθών και θα παρουσιαστούν περαιτέρω τεκμήρια και στοιχεία κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών για να δείξουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές τιμών ακόμη μεταξύ των κρατών μελών μας και σε αυτές τις διαφορές τιμών μπορεί να βρει όφελο ο καταναλωτής ε, όταν επιλέγει συνειδητά ή όταν επιλέγει online να αγοράζει. Εδώ λοιπόν σε σχέση με αυτές τις διαφορές κάνοντας καλύτερη, ε, πιο προσιτή την ε, εσωτερική αγορά στους καταναλωτές, πιο λειτουργική. Πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να διασφαλιστούν αυτά τα προτερήματα είναι με μια σωστή στοχοθετημένη, πλήρη εναρμονισμένη προσέγγιση γιατί και χωρίς τώρα να θέλω να το κάνω μια θεωρητική συζήτηση για τα ωφέλη του πλήρους εναρμονισμού, στοχοθετημένου εναρμονισμού ή ελάχιστου εναρμονισμού, επιτρέψτε μου να επαναλάβω κάποιους από τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα. Φυσικά είναι σημαντικό, όπως αρκετοί προλαλήσαντες προανέφεραν, να διασφαλίσουμε για τους καταναλωτές ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Πραγματικά δεν έχουμε άλλη επιλογή η συνθήκη απαιτεί από εμά και μας υποχρεώνει να θέσουμε επιτραπέζει και να υιοθετήσουμε προτάσεις και μέτρα τα οποία θα παρέχουν αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας. Εντάξει, Όμω είναι επίση σημαντικό να προσφέρουμε στι επιχειρήσει μας ένα ασφαλές νομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργούν και έχουν, ερχόμενοι σε επαφή με τις επιχειρήσεις αναφέρουν κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν διασυνοριακά Κάποιες από αυτές ε, δεν ε, μπορούν ή δεν έχουν κάνει τίποτα. Κάποια άλλα, κάποια άλλα θέματα οφείλονται στις παραδοσιακές διαφορές ή στις, ε, σε συνήθειες και θα έλεγα στα όσα υιοθετούνται μέσα στο πλαίσιο των παραδόσεων. Και εδώ σε σχέση με τα κέρδη τα οποία ε, μπορούν να επιτευχθούν. Όμως ένα από τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις μας λένε ότι τους δημιουργούν προβλήματα είναι ο κατακαιρματισμός, ο νομικός κατακαιρματισμός. 27 ξεχωριστά νομικά συστήματα και πλαίσια. Αυτό ίσως μπορεί να μην είναι πρόβλημα για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ε, που έχουν ε, τους νομοσυμβούλους και τις, ε, την αναγκαία τεχνογνωσία νομικά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα 27 διαφορετικά νομικά συστήματα και να διατηρήσουν τους ε, ιδίους όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με τις διαρκώς υφιστάμενες μεταβολές όμως είναι σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις ε, αυτή, αυτός ο κατακαιρματισμός. Δεν μπορούν να επομιστούν το, ε, μεγάλο, τις μεγάλες δαπάνες, το μεγάλο κόστος. Έτσι λοιπόν για τη στοχοθετημένη πλήρη, τον στοχοθετημένο πλήρη εναρμονισμό όχι μόνο είναι ε, εποφελής αλλά είναι και αναπόφευκτος αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το στόχο μας να υπάρξει μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά σε αυτό το πλαίσιο. Τούτων λεχθέντων, νομίζω ότι επίσης είναι αληθές να πει κανείς ότι προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε αυτές τις πτυχές της προστασίας καταναλωτών ε, συμβατικού δικαίου και το δικαίου συμβαλωμένων που είναι αναγκαίες πτυχές. Γι' αυτό γίνεται λόγος για στοχοθετημένη προσέγγιση και εναρμονισμό. <clears throat> Για παράδειγμα, για θέματα της, ε, όπως την ικανότητα για ε, το, ε, να συνέρχεται και να προβαίνει κανείς σε σύναψη συμβολέων. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν εντάξαμε και συνειδητά επιλέξαμε να μην συμπεριληφθούν στην πρόταση λοιπόν. Και ομολογώ και αναγνωρίζω ότι το κείμενο που έχουμε στο τραπέζι, επί τραπέζι, είναι ένα σύνθετο περίπλοκο θέμα και στην δομή και στην αρχιτεκτονική του και καμιά φορά και στην ορολογία που χρησιμοποιείται γλωσσικά. Όπως ακούσατε από την προεδρεύουσα της Σουηδική Σουηδικής Προεδρίας και η Τσεχική και η Σουηδική Προεδρία αμφότερες ε, εκπροσωπώντας τα κράτη-μέλη εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρουν αυτό το κείμενο να εξεταστεί και να γίνει καλύτερα κατανοητό. Και δεν είναι εύκολο στόχος και εύκολο έργο να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα. Αυτό το οποίο κατανοήσαμε και το είδαμε στην αντίδραση που υπήρξε σε σχέση με αρκετά επιχειρήματα που προακούστηκαν εδώ είναι το ότι κάποιες, κάποιες πρόσθετες επεξηγήσεις θα μπορούσαν να είναι επικοδομητικές. Και με αίτημα της Προεδρίας και με αίτημα των εμπλεκομένων ενδιαφερομένων πραγματικά βρισκόμαστε σε διαδικασία τώρα να ε, υπάρξει ένα επεξηγηματικό μνημόνιο, μια επεξηγηματική υποσημείωση που θα μπαίνει σε λεπτομέρειες για την αμφίδρομη δράση αυτής της πρότασης με άλλες υφιστάμενες οδηγίες και την αμφίδρομη δράση αυτής της, ε, τη διάδραση αυτής της οδηγίας με τις, εθνικ, τα, τις εθνικές διατάξεις για το δίκαιο για συμβάσεις και σύμφωνα και για επεξήγηση σε ευρύτερο πλαίσιο του εύρους αυτής της πρότασης του πεδίου εφαρμογή σε εύρος, για παράδειγμα, στο οποίο θα εφαρμόζεται όσον αφορά, για παράδειγμα, τις ε, μεταφορές, υπηρεσίε για τι μεταφορέ, ε, κοινωνικέ υπηρεσίε κτλ. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το σημείωμα για να υπάρξει αποσαφήνιση αρκετών θεμάτων που προαναφέρθηκαν σήμερα. Μια και πιέζει ο χρόνο, Πρόεδρε, δεν θα επισέλθω σε άλλε λεπτομέρειε, ε, δεν θα απαντήσω λεπτομέρω σε όλε τι παρεμβάσει και όλα τα θέματα. Τώρα, το άλλο θέμα στο οποίο βρισκόμαστε καθοδόν να προετοιμάσουμε και που ελπίζουμε και πάλι ότι θα ανταποκρίνεται σε έναν αριθμό ετοιμάτων που διατυπώθηκαν από αξιότιμους ευρωβουλευτές. Είναι ένας κατάλογος, ένας πίνακας που θα καταδεικνύει όσο σαφέστερα γίνεται με βάση τις πληροφορίες που έχουμε την διάδραση και την αμφίδρομη επιρροή που οι όροι αυτής της πρότασης θα συνεπάγονται σε σχέση με υφιστάμενες διατάξεις και, κανόνες, και κανόνες για την προστασία των, των καταναλωτών στα κράτη-μέλη. Προσπαθήσαμε έτσι, για παράδειγμα, να εντοπίσουμε και ταυτοποιήσουμε <clears throat> σε ποιες περιπτώσεις θα υπήρχε κάποια μεταβολή στο επίπεδο προστασίας ή της φύσης στην προστασία αν ε, θα υιοθετεί το χωρίς αλλοιώσεις, χωρίς αλλαγές αυτή η πρόταση από πλευρά των κρατών μελών. Και νομίζουμε ότι όλα αυτά θα δείξουν, όπως η κυρία Βάιλερ είπε, ότι θα ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη υπερβολή να πει κανεί ότι αυτή η πρόταση θα μείωνε, θα υποβάθμιζε το επίπεδο προστασία των καταναλωτών στι ε, χώρε μέλη μα. Φυσικά αληθεύει ότι αν προχωρήσουμε σε ένα πλήρη εναρμονισμό, έστω και στοχοθετημένο, αυτό θα σημαίνει ότι κάποια κράτη-μέλη θα χρειάζεται, θα πρέπει να τροποποιήσουν να αλλάξουν το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε αυτά σήμερα. Όμως εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η επίπτωση, η αξιολόγηση επίπτωσης της ε, πρόταση συνολικά θα είναι τέτοια αξιολόγηση, τέτοια αποτίμηση που την ενιαία εσωτερική αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ε, εξεταζόμενες θα βελτιώσει τα πράγματα και θα βελτιώσει και την προστασία των καταναλωτών. Πρέπει να πω ότι για την συζήτηση μέσα στους κόλπους των ομάδων εργασιών του Συμβουλίου υπάρχει εξέταση των λεπτομεριών για το επίπεδο προστασίας. Υπάρχει εξέταση λοιπόν και ε, αποτιμούμε θέματα τα οποία πρέπει να ε, βελτιωθούν για παράδειγμα σε σχέση με, την, με τις αποζημιώσεις, σε σχέση με επισκευές, σε σχέση με την αντικατάσταση ε, και παραμένει η πρωτοβουλία στους ε, εμπορευομένους ε, να επιλέξουν ποια θα είναι η αποζημίωση ή ο τρόπος με τον οποίο θα αποζημιωθούν ε, οι καταναλωτές. Και πιστεύουμε ότι αντισταθμίζεται πλήρως η σημερινή κατάσταση και η εμπορική πραγματικότητα αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο συζητείται και έχει συζητηθεί ευρέω από πλευρά των κρατών μελών και έχει συζητηθεί και εδώ σίγουρα για την διάρκεια της εγγύησης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκ του εξετάζεται πολύ προσεκτικά από τους εκπροσώπους εκπροσώπου των εθνικών κυβερνήσεων και είναι κάτι που σίγουρα χωρίς αμφιβολία και εσείς πιστεύω ότι θα επικεντρωθείτε σε αυτό όταν θα στρέψετε την προσοχή σας στις λεπτομέρειες, στα λεπτομερή θέματα αυτής της πρότασης. Αρκετά μέλη έκαναν λόγο για την ανάγκη να επιτευχθεί μια σωστή ισορροπία και θα έλεγα ότι κατανοούμε και συμμεριζόμαστε κιόλα. σίγουρα προσυπογράφουμε το γεγονός ότι Χρειάζεται, πρέπει να επιτευχθεί αυτή η σωστή ισορροπία. Η πρόταση επιτραπέζη, ε, η πρόταση που παρουσιάστηκε την Επιτροπή περίπου πριν από ένα χρόνο, έδινε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε ως αποτίμηση για αυτή την επίτευξη αυτής της ισορροπίας. Είναι σαφές λοιπόν ότι ως μέρος της νομοθετικής ε, διεργασίας και άλλες απόψεις θα διατυπωθούν για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, για το πώς μπορούμε ταυτόχρονα να προστατεύουμε με τον καλύτερο τρόπο τους καταναλωτές αλλά και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τα ωφέλη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Φυσικά η πρόταση δεν είναι κάτι το θέσφατο, το αναλύωτο ως ε, έργο, α, μήνυμα θεού ή θεολογικό. Φυσικά μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις και προσαρμογές και προσβλέπουμε στη συζήτηση αυτών των θεμάτων με την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή στο μέλλον, στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Ε, Mrs. Minor, Jackie, um, Λοιπόν, εφόσον έχουμε συνεργαστεί πολύ καιρό, σας ευχαριστώ ε, για τα ευγενή σας σχόλια και ε, επίσης για μια πολύ σαφή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που έθιξε τα περισσότερα θέματα. Μας ενθαρρύνει ότι ήδη έχετε απαντήσει σε θέματα που θίξαμε και στο Συμβούλιο και ε, χαιρετίζουμε την περαιτέρω πληροφόρηση για τις επιπτώσεις αυτής της προτάσεως, ιδίως όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ νομοθεσίας και άλλων θεμάτων. Και επίσης ε, το πίνακα τον οποίο είχαμε ζητήσει και στο παρελθόν υπό την Προεδρία της κυρίας Μακάρθη. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ χρήσιμο που είχαμε μία τόσο ευρία ανταλλαγή απόψεων και για να ολοκληρώσω σαν πρόεδρος θα ήθελα να σας πω ότι παρουσιάζοντας ε, ε, πώς ο πρόεδρος και οι συντονιστές που το συζήτησαν εκτενώς εχθές θέλουν να προχωρήσουν είναι η λήψη του, της βασικής απόφασης του καθορισμού του εισηγητή ε, και θα ε, το σκεφτούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες θα αποφασίσουμε στο Στρασβούργο δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει άσπρος καπνός πάνω από την αίθουσα σας στην περίπτωση του Πάπα αλλά εν πάση περιπτώσει, ε, θέλω να πω ότι από πλευράς της ποιότητας της συζητήσεως ε, σήμερα ε, θα υπάρξουν πολλοί υποψήφοι για το θέμα αυτό και θα έχουν δυσκολία οι συντονιστές να επιλέξουν τον τελικό εισηγήτη. Αλλά πιστεύω ότι ο εισηγητής, οι σκιώδεις θα εμπλακούν αλλά και όλοι θα μπορείτε να συμβάλλετε στις συζητήσεις αυτού του υψηλού επίπεδου σαν, όπως είχαμε σήμερα για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε την έκθεση αυτή. Το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε με τους συντονιστές και ακόμη πρέπει ε, να ε, υιοθετηθεί με την ολοκλήρωση του καθορισμού του εισηγητή είναι ότι θα ήταν καλό κάποια στιγμή στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής να υπάρξει ε, μια άλλη ακρόαση ή ένα άλλο εργαστήριο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει καλύτερα ορισμένα από αυτά τα θέματα, να ακούσουμε από το Συμβούλιο πώς προχωρούν τα θέματα αυτά, να μας πούν επίσης τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια των κρατών μελών πώς επεξεργάζονται το θέμα αυτό, διότι είχαμε μία πολύ επιτυχή ακρόαση με τους βουλευτές των ε, ε, κοινοβουλίων των Κρατών Μελών στην προηγούμενη θητεία και λάβατε ε, ηλεκτρονικά αυτή την έκθεση από τη Βουλή των Λόρδων και ο πρόεδρος της Επιτροπής με τα χαρά θα το παρουσιάσει και διεζώσεις και όσοι που από εσά ενδιαφέρονται για τα εθνικά τους κοινοβούλια ίσως ε, θα πρέπει να ζητήσετε από ε, είτε προηγούμενο προηγούμενους ευρωβουλευτές είτε βουλευτές ε, που ασχολούνται με το θέμα στο Εθνικό Κοινοβούλιο να μας ε, ε, μιλήσουν για αυτό το θέμα εδώ. Είναι βασικό για την νομοθεσία. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις και με τις οργανώσεις των καταναλωτών και σε γενικές γραμμές και υπό την αίρεση ότι θα πρέπει να καθοριστεί η συγητής. Ελπίζω ότι θα υπάρξει μία ακρόαση σε μία μεγαλύτερη αίθουσα διότι θα υπάρχει αθρώα συμμετοχή ενδιαφερομένων και θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του αποφασίσουμε. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Αυτό κλείνει το συγκεκριμένο θέμα και τέλος το επόμενο θέμα μας έχει επίσης ε, σχέση με θέματα τα οποία έχουν μεταφερθεί από την προηγούμενη θητεία. Θα δώσω την ε, δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να φύγουν. Uh, we'll just have κάνουμε μία σύντομη, ένα σύντομο διάλειμμα ε, για να μπορέσουν ε, να αποχωρήσουν ε, όσοι το επιθυμούν. Could Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω όσους θέλουν να βγουν ε, να το πράξουν και ε, να έχουμε λίγο ησυχία στην αίθουσα, κατά τρόπον ώστε να ολοκληρώσετε τις συζητήσεις σας εσείς έξω και εμείς να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουμε στην ε, Επιτροπή είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο δεν είχαμε καθορίσει εισηγητή, άρα είναι νέο θέμα στην προηγούμενη θητεία εννοώ και θέλω να δώσω τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, να μας παρουσιάσει μια επισκόπηση της προτάσεως, διότι είναι μια πρόταση για να καταργήσει, να ανακαλέσει τις οδηγίες για τη μετρολογία, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε το κοινοτικό κεκτημένο. Ε, πολλά από τα θέματα αυτά είναι πολύ παλιά, ανέρχονται στο 1971 και θα θυμάστε ότι ο εχθές το ανέφερε ο Επίτροπος Φερχόιγγεν σαν μέρος της εργασίας του και αυτός θέλει να στηρίξει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ο κύριος Χάνικομπ είναι εδώ, ο, οποίος έχει έρθει επανειλημμένος στην Επιτροπή μας, οπότε κύριε Χάνικομπ, μπορώ να σας σας ζητήσω να παρουσιάσετε την πρόταση αυτή, να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται και μετά να προτείνω στα μέλη της Επιτροπής να κάνουν ερωτήσεις ε, και να σχολιάσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή θέλει οκτώ παροχημένες οδηγίες να απαλληφθούν σε σχέση με μετρολογικά μέτρα και μετρολογικά μέτρα που είτε δεν προχωρούν τεχνολογικά επειδή πρόκειται για τεχνολογίες ειδηφιστάμενες σε σχέση με μέτρα σταθμά βάρη ή γίνονται ανεδαφικές επειδή υπάρχει νέα τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί πλέον. Παραδείγματα είναι αρκόμετρα και ε, πιεσόμετρα Παρακαλώ, οι συζητήσεις εκτός αίθουσας, εκτός αιθούσης, εντάξει. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον ομιλητή αν κάνετε θόρυβο. Λοιπόν, λυπάμαι που σας διέκοψα, δεν σας ακούγαμε όμω καθαρά. Μπορείτε να συνεχίσετε. Παρακαλώ. Ο η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να απαλληφθούν ήδη οκτώ ανεδαφικές ε, παροχημένες οδηγίες που επί μεγάλο χρονικό διάστημα ίσιαν όπω είπε ο Πρόεδρος αφαιρούν ε, μια μικρή αγορά ε, μέσων και εργαλείων που σταδιακά καθίστανται παροχημένα ή που δεν μπορούν τεχνολογικά να προχωρήσουν ε, σε σχέση για παράδειγμα με την μέτρηση βαρών. Για όλα αυτά τα μέτρα υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές διαθέσιμες αν θα ήθελαν τα κράτη-μέλη να συνεχίζουν να ρυθμίζουν αυτόν τον τομέα, δεν υφίσταται πρόβλημα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά την ίδια νομοθεσία, την κείμενη νομοθεσία. Θα υπήρχαν κάποιες μικρές ε, ελάσσονο σημασία αλλαγέ σε σχέση με κάποια θέματα. Αυτέ όμω οι αλλαγέ, αν διατυπωθούν σωστά και υπό την αρχή τη αμοιβαία αναγνώριση, δεν θα έθεταν προβλήματα, δεν θα δημιουργούσαν προβλήματα. Βρίσκονται χιλιάδε προϊόντα στι αγορέ που καλύπτονται ακριβώ από τη διαδικασία τη αμοιβαία αναγνώριση, όπου βασίζονται εθνικέ προδιαγραφέ δικαίου στι διεθνεί προδιαγραφέ. Αυτή θα ήταν η οδό για την κάλυψη των θεμάτων αυτών των οδηγιών στο μέλλον, αν θα υπήρχε κάποια προσφυγή η αντίρρηση. Στη συνέχεια υπάρχουν και άλλα νέα μέσα τεχνολογικά προηγμένης μορφής όπως για παράδειγμα πιεσόμετρα που αυτή τη στιγμή δεν έχουν εναρμονιστεί σε κανένα επίπεδο. Εκεί κάποια κράτη-μέλη μπορεί να έχουν ρυθμίσει κάποια πράγματα. Μπορούν να το κάνουν αυτό υπό και την παλαιά προσέγγιση. Η παλαιά διαδικασία τι λέει. Λέει ότι μέσα και εργαλεία τα οποία ανταποκρίνονται σε αυτή την οδηγία πρέπει να γίνονται δεκτά από τα κράτη-μέλη. Αλλά τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν και διαφορετικά πλαίσια, μπορούν να έχουν για παράδειγμα διατάξει για διαφορετικά μέσα και εργαλεία. Για αυτά τα εργαλεία και μέσα το ερώτημα είναι είναι προσκόμματα και εμπόδια στο, εμπόρευ, στο εμπόριο. Το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά σε βάθος αξιολογήθηκε ότι δεν υπάρχουν προσκόμματα και φραγμοί στο εμπόριο. Υπήρξε διαβούλευση. Κανεί στη δημόσια αυτή διαβούλευση δεν ανέφερε ότι υπάρχουν προσκόμματα και φραγμοί στο εμπόριο. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη την άποψή του. Κανένα κράτο μέλο δεν ανέφερε προσκόμματα και εμπόδια στο εμπόριο. Λοιπόν, για τα τεχνολογικά πιο προηγμένα μέσα, τα οποία ταχαίω υποκαθιστούν τώρα τα ανεδαφικά και παροχημένα τεχνολογικά, δεν υπάρχουν προσκόμματα ή φραγμοί στο εμπόριο καθότι γνωρίζουμε πλέον. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν προσκόμματα ή φραγμοί στο εμπόριο, τίθεται το ερώτημα, θα πρέπει να, να υπάρξει εναρμονισμός, για ποιο λόγο και στόχο. Λειτουργεί από ό,τι φαίνεται σωστά η διαδικασία τη αμοιβαία αναγνώρισης. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα όσον αφορά την εμπορία το εμπόριο και λαμβάνοντας αυτά υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι βασιζόμενη στην μελέτη επιπτώσεων, αξιολόγηση επιπτώσεων, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα σημαντικός λόγος για να νομοθετήσουμε ξεχωριστά κάποια νέα προσέγγιση δηλαδή. Και γι' αυτό καταλήγουμε στη διαδικασία απάλληψης, ε, κατάργησης αυτών των οκτώ παλαιών, πεπαλαιωμένων πλέον οδηγιών. Είχαμε κάποιες διαφορετικές απόψει που ακούστηκαν στο Συμβούλιο και γι' αυτό τον λόγο είπαμε προτείναμε στα κράτη-μέλη γιατί σε σχέση με οποιαδήποτε νέα στοιχεία υπήρχαν όσον αφορά φραγμού ή εμπόδια στο εμπόριο πριν από τον 10 Σεπτεμβρίου, αν μπορείτε να υποβάλλετε κάποιες ε, τέτοιες, ε, κάποια τέτοια στοιχεία και αν υπάρχει λόγο να επανέλθουμε στο θέμα, ε, στο θέμα αυτό, θα έχουμε την μελέτη επιπτώσεων. Αυτή είναι η κατάσταση ω τώρα. Περιμένουμε αυτό και θα είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι να ενημερώσουμε εσά και από πλευρά Συμβουλίου να υπάρξουν οι αναγκαίε επαφέ πριν από τα τέλη του μήνα. Για μας λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Είπαμε και αναφέραμε σε σχέση με την προηγούμενη Ευρωβουλή στα μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στο παρελθόν ότι δεδομένων των διακοιμάσεων και διαφορών σε σχέση με τις απόψεις στο Συμβούλιο για το αν θα έπρεπε να διατηρηθούν ή όχι αυτές οι ε, διατάξεις, στο τέλος υπήρξε πλειοψηφία για την κατάργησή τους. Αλλά υπάρχουν και ε, ε, ας το πω έτσι, αναχαιτιστικές ε, μειοψηφίες όσον αφορά την απάλληψη κατάργηση. Υπάρχει λοιπόν ένα μείγμα, ας το πω έτσι, αυτή τη στιγμή. Το θέμα θα είναι προσκόμματα εμπόδια στο εμπόριο. Θα είναι σκόπιμο να δούμε, να αναμείνουμε να δούμε θα υπάρξουν τέτοια επιχειρήματα που θα επικαλεστούν κάποιοι. Είπαμε στην προηγούμενη Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών ότι θα μπορούσε σε σχέση με το Συμβούλιο το Κοινοβούλιο να ζητήσει να υπάρξει επανεξέταση είτε με βέλτιστη νομοθεσία είτε με προσφυγή εναντί αυτών. Αυτό παραμένει ανοιχτή θέση ακόμα για μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος για τις πληροφορίες σας. Σαφώς καταδείξατε ότι αποδεικνύεται ότι η απλούστευση ε, είναι σημαντικό θέμα για την ε, κατάργηση ε, ανεδαφικών διατάξεων και ότι υπάρχουν ε, βαθύτερες ε, ενδείξεις ή επιπτώσεις. Η κυρία Κέπα θέλησε να παρέμβει, άλλοι θέλουν. Λοιπόν, παρακαλώ. Η κυρία Γκέπαρτ, πρέπει να ομολογήσω ότι με το θέμα αυτό δεν έχω εξοικειωθεί ιδιαίτερα στο παρελθόν και γι' αυτό δεν μπορώ να αξιολογήσω αν είναι σωστό ή λάθο αυτέ οι οδηγίε να καταργηθούν ή όχι. Αυτό όμω το οποίο θα με ενδιαφέρει πρέπει να πω είναι αν Πράγματι είναι τόσο σαφή τα πράγματα ότι πρέπει να καταργηθούν ποιοι λόγοι πραγματικά, ποια κράτη-μέλη έχουν ποιους λόγους αυτές τις οδηγίες να μην θέλουν να τις καταργήσουν. Αν μπορείτε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες εσείς για αυτά τα κράτη-μέλη θα ήταν σημαντικό για τη δουλειά μας, για μας. Διότι φυσικά ως Ευρωβουλή θέλουμε να υπάρξει απλούστευση, να εξαπλουστευτούν τα, τα πράγματα. Αν υπάρχει όμως ένα πρόβλημα για το οποίο δεν γνωρίζουμε, πρέπει να το γνωρίζουμε προτού λάβουμε απόφαση ως Ευρωβουλή. Αυτό θα ήταν το ελάχιστο που θα έπρεπε να ξέρουμε. Γιατί κάποια κράτη-μέλη, ποια κρατη και ποιο ποιου λόγου έχουν και προβλήματα έχουν για την κατάργηση αυτών των οκτώ οδηγιών. Ευχαριστώ. Uh, Άλλος που θέλει να παρέμβει. Εσείς κυρία Ρούλε παρακαλώ. Ήθελα και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου σε αυτό. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου. Θα έρθουν οι απαντήσεις μέχρι τότε των κρατών μελών. Πού βλέπουν να υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα δηλαδή. Και θα πρέπει το χρονοδιάγραμμα εργασιών μας να το διαμορφώσουμε έτσι ώστε να ενταχθεί αυτή η ημερομηνία, να ξέρουμε ευθύ εξ αρχής ποιες επιφυλάξεις υπάρχουν. Κατά τα άλλα δεν βλέπω να υπάρχει άλλο πρόβλημα. Και για τις παρατηρήσεις ε, όσον αφορά και το δικό μας χρονοδιάγραμμα, σε αυτό ήθελα να αναφερθώ. Άλλος παρακαλώ. Και κάποια σχόλια από πλευρά μου. Συμφωνώ και με τις δύο προλαλήσασες. Αλλά και ένα επιπλέον σημείο παρατήρηση. Θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτής της οδηγίας ε, το κύριο κυριότερο θέμα είναι οι λόγοι για αυτή την κατάργηση αυτών των ε, οδηγιών δεν είναι δηλαδή το να πει κανείς απλά και μόνο το ναι ή όχι και ο, λόγο, η πρότασή μου θα ήταν ευθυγραμμιζόμενος με τις άλλες προτάσεις που διατυπώθηκαν οποιοδήποτε θα αναφερθεί ως εισηγητής, θα διορθεί ως εισηγητής αποκοινούμε εσάς ε, και να μας δώσει μια αξιολόγηση αυτού του χαρτοφυλακίου, αυτού του θέματος να αποκαλυφθούν οι λόγοι που ε, οδηγούν στην κατάργηση, στην εξάλληψη αυτών των οδηγιών και νομίζω ότι θα μπορούσαμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα να το εντάξουμε αυτό ως προθεσμία, όπως είπε η κυρία Ρούλε και η κυρία Γκέπχαντ, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου να το κάνουμε αυτό, να καλέσουμε δηλαδή το Συμβούλιο να παραστεί και να σχολιαστεί το θέμα από το Συμβούλιο σχετικά. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να ζητήσω, να ρωτήσω ε, τον κύριο Χάνεκο υπό το προσωπικό πρίσμα μου είναι η διάδραση μεταξύ αυτής της πρότασης και η διαδικασία αμοιβέ αναγνώρισης ε, που τώρα εντάσσεται στο ε, πλαίσιο των αγαθών για αμοιβή αναγνώριση και για την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία ότι είναι σαφές ότι τα περισσότερα από αυτά καλύπτονται από διεθνείς προδιαγραφές με τον ένα ή άλλο τρόπο και αυτό θα υποκαθιστούσε, θα, ήταν, αντικαθιστούσε. Η νέα τεχνολογία δηλαδή ουσιαστικά θα καλυπτόταν από τις διεθνείς προδιαγραφές που ε, συντάσσονται και ισχύουν από φορείς ε, και όργανα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης αυτά θα αναγνωριζόντουσαν από τα κρατημέλη και διαρωτώ με αν και αυτό είναι μια πτυχή που θα έπρεπε να εξετάσουμε πιο καταλεπτός ε, ώστε να υπάρξει η εξέταση αυτού σε σχέση με τη μελέτη επιπτώσεων. Αυτές είναι οι δικές μου παρατηρήσεις. Διαρωτώ με, θα θέλετε να μας δώσετε κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις που να επιβεβαιώνουν και να υπαριθεύουν ότι θα είσαστε εσείς πρόθυμοι να συζητήσετε τη μελέτη και την εξέταση επιπτώσεων με αυτά τα στοιχεία και να μας δοθεί μια ε, έγκαιρη απάντηση από το Συμβούλιο σε σχέση με την ημερομηνία της 30 Σεπτεμβρίου. Συμφωνούμε, Πρόεδρε, απόλυτα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να, σας, να το συζητήσουμε, να δούμε την μελέτη των επιπτώσεων λεπτομερώς και να δούμε, να λάβουμε υπόψη μας και τις νέες πληροφορίες που θα μπορούσαν να συλλεχθούν εφόσον τα κράτη-μέλη μας πούνε τι συμβαίνει, τι ισχύει και μετά θα ήταν σκόπιμο και το Συμβούλιο να είναι παρόν και να εξηγήσει τι ισχύει για τα κράτη-μέλη. Τώρα, επί της ουσίας, συμφωνούμε απόλυτα ότι η διεθνής προτυποποίηση, αν θέλετε, η τυποποίηση, είναι αυτό το οποίο θέλουμε και το οποίο θα έχουμε σαν κατευθυντήρια γραμμή. Θα περιμένουμε και κάποια ε, κατεύθυνση να μας δώσει και ο ΠΟΕ και θα δούμε ποια είναι η διεθνή εικόνα όσον αφορά τα, την τυποποίηση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ε πρότυπα ISO που ήδη υπάρχουν. ισχύουν αυτά για διάφορα προϊόντα ε, που ανα, και αναγνωρίζονται από την ε, από τους κανονισμούς ε, της γεωργίας, στον τομέα της γεωργίας. Υπάρχουν, ε, επομένως, υπάρχει επομένως ε, νομοθεσία την οποία την παρακολουθεί και η Γενική Διεύθυνση της Γεωργίας. Τυποποίηση με βάση τους διεθνείς κανονισμούς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που βλέπουμε τον νέο κόσμο, αν θέλετε, να εισέρχεται. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να προσθέσουμε και, άλλη μια, και άλλο ένα κανονισμό. Ε, τώρα βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε σαφείς ε, ε, ανάγκες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βέβαια και το κόστος το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί εάν και εφόσον δεν υπάρχει εναρμόνιση των προτύπων. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρέπει να δούμε την κατάσταση γενικότερα. Πάντως, έτσι όπως έχουν τα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πιστώσεις στην μελέτη επιπτώσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο χρήσιμη εξήγηση και γιατί ακριβώς ε, επαναφέρεται αυτή τη ε, διαδικασία. Οι συντονιστές ε, θα το μελετήσουν και ο συντονιστή θα προχωρήσει ούτω ή άλλω. Εδώ ολοκληρώνονται οι εργασίε μας σήμερα το πρωί, λίγο νωρίτερα από ότι προγραμματίζαμε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να επιστρέψετε στις 3 ακριβώς. Θα υποδεχθούμε τον Σουηδό Υπουργό Εμπορίου που θα μιλήσει για θέματα που αφορούν την εσωτερική αγορά. Σας εύχομαι είναι η Υπουργός Εύα Μπέρλινγκ. Σας εύχομαι καλή όρεξη και θα τα πούμε στις 3 η ώρα ακριβώς.